Είστε ε, της άποψης ότι με ή χωρίς τη συμφωνία θα μπορούν να ασκήσουν περισσότερη επιρροή. Πρόεδρος, μπορείτε να απαντήσετε παρακαλώ με 30 δευτερόλεπτα. Μπορώ να απαντήσω αγγλικά, αν μου επιτρέπετε. Κοιτάξτε, βλέπουμε ότι η συμφωνία δεν βοήθησε, δεν έγινε τίποτα σε αυτή τη φάση, διότι από ό,τι φαίνεται οι διαπραγματεύσεις δεν κατευθύνθηκαν σωστά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ακολουθήσουμε αυτά που εγκρίναμε και εγκρίναμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να προωθήσουμε για μεταρρυθμίσεις και αυτά που επιθυμούμε. Όπως σας είπα, τώρα δίνουμε ελευκό επιταγή όσον αφορά το εμποριό μας. Διότι αυτοί δεν έκαναν τίποτα από αυτά που θέλαμε να κάνουν και μας είχαν υποσχεθεί. Σας ευχαριστώ και τώρα στον Φιντάντσεκ, το για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η συμφωνία αυτή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ έχει όπως πάντα επίμαχες απόψεις. Υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάποιες ε, ε, σημαντικές παραχωρήσεις για τις ε, επιχειρήσεις μας και μεγάλη προστασία για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Αλλά υπάρχουν προβλήματα όπως για ένα πολύ σημαντικό τομέα της γεωργικής παραγωγής, όπως για παράδειγμα του ρυζιού. Η παραγωγή ρυζιού τη Ιταλία. Ε, είναι ε, προβληματική λόγω των συμφωνιών με την Καμπότζη και άλλες χώρες και σήμερα στις μέρες μας έχουμε μια είδηση για εμπορικές σχέσεις με την Καμπότζη στην οποία δεν θα συμπεριληφθεί και το ρύζι στη συμφωνία. Είναι προφανώς λοιπόν ότι η διείσδυση στην αγορά και άλλων ποσοστώσεων ε, ρυζιού από το Βιετνάμ σε πολύ χαμηλές τιμές μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα έναν τομέα ο οποίος ήδη έχει υποστεί μεγάλη ζημία. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε το Ιταλικό και Ευρωπαϊκό ρύζι και εγώ δεν θα προσαπογράψω τέτοιε συμφωνίε μέχρι να γίνει αυτό. Κυρία Σιμακοπούλου, ένα λεπτό. Thank you, Madam President. Στηρίζουμε τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Ευρωπαϊκή Ένωση και Βιετνάμ, γιατί είναι μια πολύ καλή συμφωνία η οποία έχει οικονομικά ωφέλη για όλου. Με τη σταδιακή κατάργηση σχεδόν όλων των δασμών, με την άρση των δασμολογικών ποσοστώσεων, ανοίγοντα τι αγορέ στου παρόχου υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και δίνοντας πρόσβαση στους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων. η συμφωνία έχει ωφέλη για πολλά κράτη μέλη μεταξύ των οποίων και της δικής μου χώρας της ελλάδας όπου θα βοηθήσει στις εξαγωγές φαρμακευτικών ειδών και αγροτικών προϊόντων εξασφαλίζοντας την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων σημαντικών ελληνικών προϊόντων όπως είναι η φέτα και το ούζο. επιπλέον η συμφωνία θα θωρακίσει τα εργατικά δικαιώματα θα ενισχύσει τη δημοκρατία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα συμβάλλει στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. οπότε στην εποχή των εμπορικών πολέμων έχει και μια συμβολική αξία καταδεικνύει ότι η ευρωπαϊκή ένωση επιμένει σε ένα πολυμερές σύστημα ελεύθερου εμπορίου βασισμένο σε δίκαιους κανόνες που συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της ενωμένης ΕΕ. ευρώπης. σας καλώ να την υπερψηφίσουμε. ευχαριστώ. πολύ. λεπτό. Er Ευχαριστώ πολύ. Σε μια εποχή που η ελευθερία και η συνεργασία ε, στέλνεται από παλιούς φίλους, ε, καλό θα ήταν να ανοίξουμε νέες αγορές, ε, να κάνουμε νέα ανοίγματα. Βέβαια θα πρέπει το εμπόριο να βασίζεται και σε κανόνες, σε αρχές. Θα πρέπει να στηρίξουμε αυτή τη συμφωνία. Είναι η πληρέστερη συμφωνία που έχει συναυτεί ποτέ μεταξύ μιας αναπτυσσόμενης χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Βιετνάμ έχει εγκρίνει ήδη έξι συμβάσεις ε, της ε, Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ε, και υπάρχουν πραγματικά διαπραγματεύσεις που μπορεί να οδηγήσουν και σε την ελευθερία του συνεταιρίζεστε για 95 εκατομμύρια ανθρώπου. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν δεν είχαμε τίνει εμείς χείρα στην χώρα αυτή και σίγουρα ο στόχος δεν είναι ε, τελειομανία, ε, αλλά συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Βίντσικ, ένα λεπτό είναι επόμενη μιλήτρια. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ιστορία έχει δείξει πως το εμπόριο και οι ανοιχτές αγορές δημιουργούν ευημερία, ασφάλεια. Είμαι από μια χώρα ε, που έχει ε, πολλές ε, εξαγωγές και κάθε δεύτερη θέση εργασίας άμεσα ή έμεσα σχετίζεται με τις εξαγωγές. Και θεωρώ ότι αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε το κοινωνικό μας σύστημα δεν μπορούμε να το πετύχουμε χωρίς εξαγωγές. Ε, πράγματι είναι πολύ σημαντικές οι σχέσει και οι συμφωνίες αυτές ε, με το ε, χώρα του Βιετνάμ που είναι μια σοσιαλιστική αναδυόμενη χώρα και ανοίγει νέες δυνατότητες. Σίγουρα πρέπει βέβαια η χώρα να εφαρμόσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και υπάρχει και η πολιτική διάσταση, δηλαδή ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρέπει να υπάρχει ο μηχανισμός αξιολόγησης και επιβολής κυρώσεων. Αυτό είναι θετικό. Και κάτι άλλο θετικό, το που και ο κύριο προηγουμένω είναι αυτά τα εργασιακά πρότυπα ε, που θα πρέπει να έχουν εγκριθεί οριστικά μέχρι το 2030 οικονομική ε, επιτυχία της Ευρώπης ε, ίσως ε, να μην ενδιαφέρει τόσο άλλους, όμως νομίζω ότι πρέπει εμείς να συνεχίσουμε, γιατί και από πολιτική πλευράς έχει μεγάλη σημασία με τέτοιου είδους συμφωνίες. Ευχαριστώ λίγο Σκέλη για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε Χόγκαν, και κύριε Σιγητά, κύριε Μπυρσουά και οι υπόλοιποι, θα επισημάνατε πάρα πολλά από τα ωφέλη αυτής της ε, συμφωνίας και για το Βιετνάμ αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ούτως ή άλλως οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να είναι συμφωνίες από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι όλοι. Και ως ε, μόνιμος συγητής για την περιοχή του ΑΣΕΑΝ και η συγητής ε, για το ΕΛΚ, σκιώδη συγητής για τη Σιγκαπούρη, καλωσορίζω την συμφωνία με το Βιετνάμ. Είναι η πρώτη πλήρη συμφωνία που συνάπτουμε με μια αναπτυσσόμενη χώρα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ε, συμφωνία με αναπτυγμένη οικονομία είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι θετικό λοιπόν το μήνυμα ότι συνάπτουμε συμφωνίες με αναπτυσσόμενες χώρες όπως το Βιετνάμ. Για όσους είναι αντίθετοι θα είχα να πω ότι πολλά από τα προβλήματα που έχετε ε, θα βελτιωθούν αν ε, ε, εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Ε, η απάντηση είναι όχι. Υπάρχουν τεράστιες βελτιώσεις οι οποίες προέκυψαν ήδη και από τι διαπραγματεύσεις και θα συνεχιστούν ε, κατά την εφαρμογή της συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Χόγκεν, η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορία με το Βιετνάμ αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και εκτό και εντό Ευρώπη. Εκτό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι η μεγάλη εμπορική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποδεικνύει ότι παρά τα όσα κάνουν οι λαϊκιστέ για να ε, υψώσουν ε, ε, δασμολογικού φραγμού και να επιβάλλουν προστατευτισμό, η Ευρώπη ηγείται του ελευθέρου εμπορία και είναι πάρα πολύ σημαντικό και εντό Ευρώπη για τι χιλιάδε οι οποίοι βλέπουν την εξαφάνιση του 75% των δασμών, μεγάλες ευκαιρίες για εμπόριο, μια νέα αγορά που ανοίγεται όταν κλείνουν άλλες. Για την Ισπανία αυτό θα είναι ουσιαστικά εποφελές για το μέσο, όπως για παράδειγμα ε, ε του τομέα του ελαιολάδου, τον τομέα του της επιτραπέζια Ελιάς ε, και των ε, πνευματιδών ποτών και του Ίνου που έχουν και προστασία γεωγραφικής ένδειξης ε, και προστασίες ονομασίας προέλευσης. Για όσους δεν τηρούν τη συμφωνία θα επαγρυπνούμε, ώστε να φροντίσουμε η συμφωνία να μην υπογραφεί για το τίποτα και όλοι οι Ευρωπαίοι και οι Ισπανοί να βγούμε κερδισμένοι από τη συμφωνία. Γι' αυτό προτείνω να υπερψηφίσουμε τη συμφωνία. Η κυρία Σόφκο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το Βιετνάμ είναι ένας πολύ σημαντικό εταίρος στην Νοτιοανατολική Ασία. Φέτος ήταν προέδρη τη ΑΣΕΑΝ και ε, είναι πολύ σημαντικό ότι προχωρούμε σε εμπορικέ σχέσει. Με αυτή τη Συμφωνία Ελευθέρω Εμπορία ξεκινάει μια νέα εποχή στη σχέση μας. Το Βιετνάμ είναι μια οικονομία που αναπτύσσεται ταχύτατα και η συμφωνία αυτή προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές ενθαρρύνουμε ε, πολιτιστικές και οικονομικές ανταλλαγές ε, και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από περιφέρεια σε περιφέρεια και σχέσεις εμπορικέ με την Νοτιοανατολική Ασία. Επίσης, ε, θα ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή προβολή στις ασιατικές αγορές. Πέραν όμως του εμπορίου και της συνεργασίας, πρέπει να έχουμε κατά νου και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα εταίρων. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση περιορίζει την μέσω της οι τοπικές αρχές πολλές φορές ε, δημεύουν περιουσίες σε χώρους λατρείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα πρέπει να πιέσει για διαθρησκευτικό διάλογο. Δεν θα πρέπει να ε, προχωρήσουμε μόνο σε ενίσχυση των οικονομικών δεσμών, αλλά και το δικαίωμα τη ανεξιθρησκεία ως ε, πολύ σημαντική πτυχή των μελλοντικών σχέσεων. Υποστηρίζω αυτή την εμπορική συμφωνία, αλλά περιμένω και πολύ στενότερη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Μπέντελε τώρα για ένα λεπτό. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, με συνάδελφοι, εγώ στηρίζω την σύναψη των συμφωνιών με το Βιετνάμ γιατί θα δημιουργήσουν και θα διατηρήσουν θέσεις εργασίας στο Βιετνάμ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια θετική εξέλιξη που δρομολογείται που θα έχει θετικές επιπτώσεις και για την κοινωνία ή θα μπορεί να έχει δυνητικά θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία. Βέβαια θα πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό νομικό πλαίσιο και ένας χώρος διαλόγου, ένας μηχανισμός ελέγχου και η ε, Επιτροπή με και από τις δύο πλευρές που θα επιβλέπει την εκτέλεση των συμφωνιών γιατί θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με το Πράσινο Σύμφωνο και το, τη Συμφωνία των Παρισίων. Έχουμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν δίνουμε μια εντλευκό εξουσιοδότηση. Υπάρχουν προϋποθέσεις και όροι. Και τώρα έχει η Κομισιόν την υποχρέωση το χρέος να δημιουργήσει ένα μοντέλο, να κάνει παράδειγμα αυτή τη συμφωνία και ελπίζω και άλλες χώρες να θελήσουν να αξιοποιήσουν την ίδια αυτή δυνατότητα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Επόμενη ομιλήτρια είναι η Σάφος Περέιρα. Για ένα λεπτό έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Βιετνάμ, πέρα από το ότι είναι εποφελή συμφωνία από πλευρά οικονομική επηρέασε ήδη τι εξελίξει, διότι υπάρχει ένα κώδικα ε, για τι εργασιακέ σχέσει στο Βιετνάμ, για τι συλλογικέ συμβάσει, ελευθερία των συνδικάτων. Όλα αυτά τα επιτεύγματα οφείλονται στη δράση μα. Δεν μπορώ να μην επισημάνω όμω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι όσον αφορά την έγκριση της σύμβασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εργασία για την κατανακαστική εργασία και για τη συμμόρφωση με τη Συμφωνία των Παρισίων, διότι δεν γνωρίζει σύνορα η αλλαγή το, του κλίματο. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μα για να δεθώσουμε την κατάσταση αφορά το κλίμα. Είναι μια συμφωνία που δείχνει πώ η πολιτική μα, η εμπορική, μπορεί να προωθήσει τι αρχέ και τι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίτροπε, συνάδελφοι, χάσαμε το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά παραμένουμε παρόλα αυτά μεγάλη εμπορική δύναμη δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω όσον αφορά το να εκφράσουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προωθήσουμε τα κοινωνικά δικαιώματα, τα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιοποικιλότητα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω 7 ε, αιτήματα για συνάδελφους που θέλουν να πάρουν το λόγο υπό τη δικασία προσοχής προσοχής του Προέδρου, συνάδελφος Ντέιλι. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις ήδη ανθούν στο Βιετνάμ. Πολύ μεγάλη αύξηση οικονομίας, ευκαιρίες, κέρδη και είναι ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε το λαό το περίπου 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Γι' αυτό είχαμε τις ε, πιέσεις από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και πιέσει που ασκήθηκαν από οργανώσει των επιχειρηματιών να μην αναβληθεί η κύρωση συμφωνία. Α μην αυταπατώμεθα το κάνουμε αυτό για το όφελο του βιετναμικού λαού. Αυτή η συμφωνία είναι για να του βγάλουμε από τη φτώχεια. Σαν κάποιο με γελίο τρόπο διατείνεται, αυτέ οι συμφωνίε κατέληξαν σε μεταφορά πλούτου από το, από νότο του κόσμου προ τη Δύση. Πονομεύονται σε απασχόληση, ανάπτυξη σε χώρε όπω είναι η Ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πει πώ θα λύσουμε τα προβλήματα, θα αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι αλαζονικό. Οι Βιετναμοί θα το δουν αυτό που οργανώνονται οι Βιετναμέζοι όπω έκαναν οι λαοί στι άλλε χώρε. Και αν είμαστε σοβαροί για τι ανησυχίε του, θα ακούσαμε τι ΜΚΟ και τα, εμπορικά, και τα συνδικάτα που μα λένε να μην κυρώσουμε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Συμφωνία Εμπορικών ε, η πολιτική συγγνώμη εμπειρικών συμφωνιών που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τα τελευταία χρόνια αποδεικνύεται ένας πολύ σημαντικός ε, παράγων για να ε, προωθήσουμε περιβαλλοντικά και κοινωνικά δικαιώματα και κυρίως θεμελιώδη δικαιώματα πολύ σημαντικό σε αυτή τη συμφωνία. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εφαρμόσει αδύνατες πολιτικές σε κάθε χρόνο χώρα και έχοντας έτσι προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες. Χαίρομαι επίσης ότι αυτή η συμφωνία λαμβάνοντας υπόψη της και ένα πιο δίκαιο εμπόριο δεν ξεχνά κανένα τομέα. Έτσι ε, δίνονται κάποια μέτρα ώστε να φροντίσουμε κάποια παραγωγή, κυρίως ε, μεταποίηση αλίας και κυρίως ε, η κονσερβοπία, θα μπορέσουν να έχουν προστασία των συμφερόντων τους και αναγνώριση των καλών πρακτικών για την, σε αντίθεση με την παράνομη λαθρέα και άνεργη ε, Αν δεν αποσύρει την κίτρινη κάρτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατεύει τις παράνομες αυτές αλληλευτικές πρακτικές. Ευχαριστώ. Αρενά είναι η επόμενη συνάδελφος. Ευχαριστώ η υπερψήφιση μια φιλελεύθερη εμπορική συμφωνία με ένα αυταρχικό κομμουνιστικό καθεστώ στο όνομα τη πράσινη ανθρωπίνων δικαιωμάτων πραγματικά είναι ε, υπερρεαλιστικό. Ξέρετε ότι είμαι από το Βέλγιο που είναι χώρα του σουρεαλισμού, όπω και ο κ. αλλά εδώ παίρνουμε πια ε, τη χρυσή σφαίρα και ο Χρυσό Φίνικα. Ε, νομίζω θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα, γιατί ο μηχανισμό επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών. Γιατί δεν καλύπτει βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί όταν πρόκειται για κοινωνικά περιβαλλοντικά δικαιώματα, δεν υπάρχει δεσμευτικό μηχανισμός με υποβολή κυρώσεων. Μία τέτοια αλλαγή είναι δυνατή, είναι εφικτή κύριε Επιτροπέ. Πρέπει να υπάρχει όμως πολιτική βούληση γι' αυτό. Εσείς ε, και εμείς ως Κοινοβούλιο νομίζω έχουμε το χρόνο να τροποποιήσουμε ε, τη συμφωνία όπω το κάναμε με το ESDS. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν κάτι πολύ καλό, ε, αγωνιστήκαμε Αλλάζοντας ε, το ESDS στο ECS κερδίσαμε, ας κάνουμε κάτι ανάλογο ώστε ε, να μπει και κεφάλαιο βιωσιμότητας δεσμευτικό με κυρώσεις. Ευχαριστώ. Ολα είναι επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Επίτροπε, μας είπατε τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν θέμα που μας ανησυχούσε για το Βιετνάμ. Πείτε με, για όνομα του Θεού, Πότε τέτοιες ανησυχίες ανθρώπινα δικαιώματα έχουν παρέμβει με τα επιχειρηματικά μα συμφέροντα. Κάνουμε, έχουμε επιχειρηματική σχέση με Σαουδική Αραβία και Ισραήλ. Αυτές οι εμπορικές συμφωνίες δεν κάνουν τίποτα για τους λαούς των περιοχών. Αποδεκατίζουν την τοπική βιομηχανία, φτωχαίνουν τους μικρού γεωργούς. Ο λαό του Βιετνάμ δεν θα ωφεληθεί από αυτό. Οι μεγάλες επιχειρήσει του Βιετνάμ θα ωφεληθούν από τη συμφωνία. Το βασικό πρόβλημα με αυτού του είδους τη συμφωνία είναι ότι εγγυάται εφαρμόσιμα δικαιώματα σε ξένους επενδυτές και τις πολυεθνικές. Και η ρήτρα περιφθής των διαφορών δεν προβλέπει κυρώσει για μη συμμόρφωση με κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Τι πιθανότητες έχει να έχουμε εμπορικέ σχέσεις ε, με αυτή τη χώρα που είναι μακριά στον πλανήτη και να είναι καλή για το περιβάλλον συμφωνία. Μηδέν. Ότι συμφωνεί με τη Συμφωνία των Παρισίων. Μηδέν μηδέν πιθανότητες να συμφωνεί με τις επιταγές. Ευχαριστώ πολύ, Κάνιας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε δεν θα έπρεπε η άγνοια να αιτιολογεί δημαγωγικά επιχειρήματα, ειλικρινά. Υπάρχει εμπόριο με το Βιετνάμ, γιατί ε, κλείνουμε τα μάτια μας στο προφανές. Μα υπάρχουν, ε, έχουμε 13 δις εισαγωγών και πάνω από 40 δις εξαγωγών, άρα υπάρχει, είναι αλήθεια. Και τι θέλουμε, απλά θέλουμε να προσαρμοστεί σε κανόνες. Ε, αυτό θέλουμε, γιατί θα, τονεί, θα τονώσει, θα ωφελήσει και τους στόχους μας ανάπτυξης, την προστασία των δικαιωμάτων, το περιβάλλον, μέλλοντος βελτιώνουμε τη συμφωνία και καλύτερο είναι να έχουμε μια συμφωνία παρά καμία συμφωνία. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο με διακηρύξεις ε, και με ακραίες ε, φιλοπεριβαλλοντικές ακραίες απόψεις. Πώς θα βελτιώσουμε με τα λόγια τη ζωή των πολιτών. Δεν θα τη βελτιώσουμε με τα λόγια. Αυτή τη συμφωνία έχουμε ένα ε, όριο, ένα πλαίσιο που δημιουργεί και κανόνε και υποχρεώσει. και εμεί έχουμε αυτό το χρέο ε, να είμαστε σε γρήγορες, να απαγρυπνούμε να εφαρμόσουμε σωστά. Αλλά ε, κρέε, εξτρεμιστικέ τέτοιε δηλώσει, όχι, γιατί το μόνο που θέλουν είναι ε, η άγρα ψήφων και όχι η βελτίωση των κοινωνικών, εργασιακών, ανθρώπινων δικαιωμάτων, η προστασία του περιβάλλοντο και καταπολέμηση της Ευχαριστώ. Ζωνκ, επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου και γι' αυτό υποστηρίζω τη σύναψη της ε, συμφωνίας. Έχω όμως κάποια ανησυχία που θα ήθελα να εκφράσω απευθυνόμενος προς τον Επίτροπο και ζητώ απάντηση. Πρέπει να υποθέσουμε ότι οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα τρόφιμα από το Βιετνάμ θα αυξηθούν. Τώρα είναι στην τέταρτη ή πέμπτη θέση. Στο μέλλον θα αυξηθεί η θέση των εισαγωμένων τροφίμων. Ερώτηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προετοιμασμένη να ελέγχει αυτά τα τρόφιμα από πλευράς ποιοτική. Δεν θα επηρεαστεί η αγορά μας τροφίμων όσον αφορά ε, το παραεμπόριο, παράνομη εισαγωγή ε, τροφίμων στην Ευρώπη που δεν θα είναι καλής ποιότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Σόλτς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ας δούμε το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Πόλεμος απελευθέρωσης, ε, ε, Βιετνάμ, ε, με πολύ βίες πτυχές και έπειτα είχαμε το μετασχηματισμό στο Βιετνάμ και υπήρξαν ε, από την ε, ηγεσία της χώρας ε, αποφάσεις για το άνοιγμα της χώρας και γι' αυτό ακριβώς αγαπητοί συνάλφοι Ζήμων Κάνιας υπάρχει τώρα αυτή η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ και θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης, ε, το περιβάλλον, ε, ε, τη ελευθερία του συνεταιριστή και γι' αυτό χαίρομαι που μπορούμε να υποστηρίξουμε επίσης τη χώρα αυτή που έχει υιοθετήσει τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Υπάρχουν όμως και κάποια κεφάλαια που μπορούν να βελτιωθούν και χαίρομαι που μπορούμε να υιοθετήσουμε υλοποιήσουμε πλέον αυτή την ε, συμφωνία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόγκαν έχει τώρα το λόγο μετά το πέρας αυτής της ανταλής απόψε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τη συμβολή του και είναι και μια ευκαιρία να ευχαριστήσω ανθρώπους που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ. Τον κύριο Λάγκε, πρόεδρο της ε, Διοργανικής Επιτροπής και όσοι συμμετείχαν στον έλεγχο αυτής της συμφωνίας και τους τέσσερις πρόεδρους των Επιτροπών που εμέσως συμμετείχαν σε αυτόν τον έλεγχο και έδωσαν την υποστήριξή τους για τη συμφωνία. Να ευχαριστήσω την πρώην Επίτροπο τη Εσίλια Μάλστρομ και τη Γενική Διεύθυνση Trade και τους υπαλλήλους για τη στερά τεράστιες προσπάθειες που έκαναν ε, πολλά χρόνια για αυτή τη συμφωνία. Όπως είπαν πολλοί από τους ομιλητές, ε, αυτές είναι, αυτή μάλλον είναι η πρώτη συμφωνία που θα ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο και ελπίζω να την εγκρίνετε, ώστε οι επιχειρήσεις μας, ιδίω οι μικρομεσαίες που αναφέρθηκαν από πολλούς από εσά, να ξεκινήσουν να απολαμβάνουν τα ωφέλη ε, αυτής της συμφωνίας και να υπάρξει ανάπτυξη. Σε χαλεπούς καιρούς για το εμπόριο είναι πολύ σημαντικό να σταλεί ένα μήνυμα ε, για τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα εμπόριο το οποίο βασίζεται σε αρχές και αξίες. Και θέλω να συμφωνήσω με πολλού από εσά ότι όντω υπάρχουν θέματα προ επίλυση και σίγουρα θα πρέπει συνεχώ να είμαστε σε εγρήγορση ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το Βιετνάμ θα τηρήσει τι δεσμεύσει του. Συμφωνώ πολύ ε, με αυτή την αίσθηση. Αλλά ε, το εμπόριο συνήθω ε, ε, συνδέεται με την πρόσβαση στην αγορά και αυτή είναι πολύ καλή συμφωνία ε, για πολλά προϊόντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Βιετνάμ αλλά αναφέρθηκαν και κάποια θέματα για τρόφιμα και πρέπει να πω ότι η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ε, απελευθερώνει όλα τα επιθετικά συμφέροντα όπω για παράδειγμα το βόλιο κρέα, τα ενοπνευματόδη, τον ίνο και την πύρα αλλά και για κάποια ευαίσθητα θέματα όπω για παράδειγμα το ρύζι, το ζαχαρότευτλο και τον τόνο σε κονσέρβα. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα για τι εμπορικέ μα συμφωνίε τα πρόσφατα χρόνια και για πρώτη φορά υπάρχει μια συμφωνία ελευθερωμποριού όπου υπάρχουν δικλείδε αλφαλίας για του κανόνε ε, προστασία προέλευση και υπάρχει και δέσμευση από πλευρά ε, Βιετνάμ για να θεωρείται ως ένας ενιαίος φορέας Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον που θα δημιουργήσει και μείωση σε πολλού μη δασμολογικούς ε, φραγμού που έχουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί προστατεύονται και πάρα πολλά προϊόντα για το, η βελτίωση της εφαρμογής ε, και της, βελτίω, της ε, ε, παρακολούθηση συμφωνία είναι πολύ σημαντικό. Ε, το Βιετνάμ έκανε πολύ σημαντικές προσπάθειες. Ε, ε, έχει αρχίσει να φροντίζει και κάποια θέματα πριν από την έναρξη εφαρμογή τη συμφωνία. Επομένω, οι πιέσει σα αποφέρουν καρπού. Επίση, υπάρχει και μια θεσμική δομή η οποία θα περιλαμβάνει όλου του ενδιαφερομένου μη κυβερνητικέ οργανώσει, την κοινωνία των πολιτών, τι επιχειρήσει και όλε τι υπηρεσίε και θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην εφαρμογή αυτή τη συμφωνία. Η εφαρμογή είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό επίση ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει και ένα ε, αρμόδιο ε, επικεφαλή για την εφαρμογή τη συμφωνία που θα καθοριστεί του επόμενου μήνε. Επίση, αναγνωρίζεται η αρχή τη ελευθερία του συνέρχεστε που θα βοηθήσει και κάποια συνδικάτα που αναφέρονται και είναι εκτό του πεδίου εφαρμογή τη γενικότερη συμφωνία για την εργασία του Βιετνάμ. Το Βιετνάμ έχει ξεκινήσει με την εφαρμογή, έχει ένα σχέδιο το οποίο θα ξεκινήσει την εφαρμογή του από 2021 πρώτη πρώτου και θα κοιτάξει να δει αν υπάρχει συνέπεια με όλα τα νομικά κείμενα και σε ποινικό και σε αστικό επίπεδο. Ε, και αν εφαρμοστούν όλα αυτά και θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται. Ε, ήταν στο ίδιο στάδιο με την εφαρμογή με την Ιαπωνία. Άρα είναι πολύ σημαντικά τα βήματα που έχουν κάνει στο Βιετνάμ. Υπάρχουν ανεξάρτητε οργανώσει τη κοινωνία πολιτών και μου έχουν δώσει και ένα πρόγραμμα δράση και χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων. Αναφέρθηκε η παιδική εργασία, μείωση από το 2012 σε 40% και επίση ε, θέλουν να εκριζώσουν την παιδική εργασία σε ένα νέο ε, σχέδιο εργασία για να καλύπτουν το διάστημα 2021-2025. Πολλοί αναφέρθηκαν στα ανθρώπινα δικαιώματα και σωστά είναι ένα τομέα στον οποίο θα πρέπει να ανησυχούμε στη σχέση μα με το Βιετνάμ. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και από πού ξεκίνησε αυτή η χώρα και να δούμε ότι όντω τα τελευταία 25 χρόνια υπήρξε τεράστια πρόοδο, ιδιαίτερα στο κοινωνικό-οικονομικό τομέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικέ ε, οι διατάξει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ε, πλήρη ή μερική αναστολή τη συμφωνία όταν υπάρχουν συστηματικέ ή πολύ σοβαρέ παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίση, υπάρχει ένα ετήσιο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μάλιστα συνεδριάζουν την επόμενη εβδομάδα στο Ανόη. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά ε, και δεν λέω και κάτι αντίθετο, αλλά χαιρόμαστε που υπάρχει μια αρχική πλατφόρμα για να έρθουμε σε επαφή με την κοινωνία του Βιετνάμ και με τι κυβερνήσει για τα θέματα αυτά. Και αυτό είναι θέμα το οποίο τονίζουν και πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσει στο Βιετνάμ. Θα ανοίξει χώρο για την κοινωνία των πολιτών. Φαίνεται ότι οι συνάδελφοι δεν έχουν ακούσει αυτέ τι δηλώσει για αυτό το τμήμα τη συμφωνία. Η συμφωνία βέβαια έχει και άμεση σχέση με του πολιτικού κρατουμένου ε, και τα άτομα ενδιαφέροντα έχουμε ένα κατάλογο ατόμων ε, ε, σημαντικού ενδιαφέροντος, το οποίο λαμβάνουμε υπόψη και αναφέρουμε στις επαφές που έχουμε σε ανώτατο επίπεδο με το Βιετνάμ συνεχώς και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα απελευθερωθούν αυτοί οι άνθρωποι, θα υποστούν μια δίκαιη δίκη, θα συναντήσουν την οικογένειά τους και θα υπάρχουν οι καλύτερες δυνατές εγκαταστάσει για αυτού του πολιτικού κρατημένου. Η Συμφωνία λοιπόν Ελευθέρου Εμπορίου και Ελευθέρου Συναλλαγών θα είναι ένα πολύ σημαντικό περιβάλλον ώστε να εξασφαλίσουμε τα θέματα αυτά. Δεν θα τα κρύψουμε κάτω από το τραπέζι, αλλά θα είναι συνεχώ στι προτεραιότητέ μα στο θεματολόγιο μα. Και φυσικά, εάν δεν υπήρχε συμφωνία, δεν θα είχε κανένα εργαλείο η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξει ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων. Εμεί θέλουμε, όπω ε, και άλλοι εταίροι που δεν ε, ε, έχουν αντίστοιχε αξίε, να υποστηρίξουμε το Βιετνάμ. Και υπάρχουν πολλά βήματα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτά τα βήματα. Το Βιετνάμ είναι μία από τι χώρε που πλήγονται περισσότερο, πλήττονται συγγνώμη, περισσότερο από την κλιματική αλλαγή και επομένω είναι πάρα πολύ σημαντικό να εφαρμόσουν τη Συμφωνία των Παρισίων, την οποία έχουν προσυπογράψει. Και ε, στο κεφάλαιο βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται ρητά η Συμφωνία. Επομένω θα πρέπει να υπάρξει συμβολή για να εξασφαλίσουν ότι όπω και σε άλλε περιοχέ του κόσμου που κάνουμε τέτοιε συμφωνίε θα τα εφαρμόσουν αυτά όπω τα υπέγραψαν και στη Συμφωνία των Παρισίων. Είναι ένα άλλο λοιπόν παράδειγμα όπου παρέχουμε το πλαίσιο για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μέσω αυτή τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου και να πιέσουμε για να εξασφαλίσουμε ότι εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά. Το Βιετνάμ επίση έχει μια εθελοντική εταιρική σχέση για ε, θέματα δασικά και την εφαρμογή του FLEGT που εφαρμόζεται από τον Ιούνιο του 2019. Και ιδιαίτερα αυτή η συμφωνία εξασφαλίζει ότι όλα τα προϊόντα ξυλία που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Βιετνάμ είναι νόμιμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ε, το Βιετνάμ είναι ε, κόμβος μεταποίησης ε, ξυλίας και από χώρε όπω η Καμπότζη και άλλες στις ασιατικέ περιοχές. Υπάρχουν λοιπόν υποχρεωτικές υποχρε... για δέουσα επιμέλεια και το Βιετνάμ φροντίζει να υπάρχει εφαρμογή του προγράμματο. υπάρχουν διάφορε άδειε για να εξασφαλίσουμε και χνηλασιμότητα. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία επιτυχία επίση είναι η δυνατότητα συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και αυτά είναι θέματα τα οποία ετέθησαν και λάβαμε απαντήσεις και θα πρέπει να συνεχίσουμε τελικά ώστε να επιτύχουμε τον τελικό μας στόχο και προορισμό. Τέλος, όσον αφορά το σύστημα των επενδύσεων και την επίλυση διαφορών, ε, λόγω των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε ε, στη συμφωνία το καλύτερο πλαίσιο προστασίας των επενδύσεων και υπάρχει ε, σύστημα επίλυσης διαφορών το οποίο αντικαθιστά τον παραδοσιακό μηχανισμό ISDS ε, και αυτό είναι αυτό το οποίο ε, επέδειξε και η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Φροντίζονται λοιπόν να συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά στη συμφωνία με το Βιετνάμ που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ορόσημο για ε, ένα δικαστήριο πολυμερών επενδύσεων. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι υπερψηφίζοντα αυτή τη συμφωνία, υποψηφίζεται μια συμφωνία που θα μας δώσει την πολιτική και θεσμική επιρροή και τις κατάλληλες δομές για να κάνουμε αλλαγέ σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασιακών δικαιωμάτων, κλιματικής αλλαγή και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων. Εάν καταψηφίσετε, ε, αφήνετε τη δυνατότητα ε, να υπάρχουν μέτρα τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα τα γνωρίσουν. Έτσι, το Βιετνάμ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετέχουν σε μια πολιτική δομή και σε μηχανισμού επιβολή που θα επιτύχουν κοινού στόχου κυρίω στους τομείς πολιτική που αναφέρθηκαν εδώ στο Κοινοβούλιο. Και ξέρω ότι πολλά από αυτά τα θέματα σα ανησυχούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουμε πλέον ένα διαρθρωμένο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Ήγηκε λοιπόν η ώρα να υπερψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία και να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει και το λαό του Βιετνάμ. Και για την ολοκλήρωση συζήτηση, το λόγο έχει ο κ. Μπουρζουά, Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητέ Πρόεδρε, συνάδελφοι, αγαπητέ Επίτροπε. Στο τέλος της συζητήσεως θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ, τους σκιώδεις εισηγητές και κυρίως ευχαριστώ τον Πρόεδρό μας, τον κύριο Λάγκερ, να ευχαριστήσω τον προκάτοχό μου, τον πρώην εισηγητή, τον Γιάνν Ζάχραντιλ. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, τον κύριο Χόγκαν, για την καλή μας συνεργασία που σωστά υπογραμμίστηκε η συμφωνία αυτή η συμφωνία για το εμπόριο και τις επενδύσεις ε, ε, είναι όπως το περιγράψατε στα συμπεράσματά σας. Και σημειώνω ότι δεσμευθήκατε σαφώς να εποπτεύετε όλες τις πτυχές που αφορούν την υλοποίηση της συμφωνίας και τη συνεχή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να βοηθηθεί το Βιετνάμ να επιδιώξει τη μεταρρυθμική του διαδικασία και να δώσουμε στη χώρα τα αναγκαία μέσα τεχνικά και οικονομικά, ούτω ώστε να πετύχει τους στόχους της. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, σας ευχαριστώ για την πολύτιμη συνεισφορά σας. Τα περισσότερα σημεία ανησυχιών που εξεφράσαν στη συζήτηση ήταν και δικές μου ανησυχίες. Όμως, πιστεύω ότι Έχουμε διασκεδάσει επαρκώς τις περισσότερες ανησυχίες στην προπαρασκευαστική μας εργασία. Πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία θα εξυπηρετήσει σαν αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόθεση θεμελιωδών αξιών και την παραγωγή πιο ισοτήμων συνθήκων για το εμπόριο. Δεσμεύτηκε το Βιετνάμ να, κάνει μια σειρά, να εφαρμόσει μια σειρά σημαντικών μέτρων και συμφωνώ με εσά κύριε Λάγκα ότι χάρη στα σαφή πολιτικά μηνύματα του Κοινοβουλίου θα γίνουν αυτά. Με τα χαράς λέγω ότι κατά τις διαπραγματεύσεις πριν από αυτή τη συζήτηση και κατά τη διάρκεια των δικών μου επαφών η βιετναμική κυβέρνηση απέδειξε ότι είναι αξιόπιστη και ότι έχει πολιτική προθυμία να ε, συμμορφωθεί με βασικά σημεία ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν σημαντικός όσον αφορά όλα αυτά. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την όλη διαδικασία όσον αφορά τις ανεξάρτητες οργανώσεις ε, που συμμετέχουν στις εγχώριες συμβουλευτικές ομάδες. Μετά την εκκύρωση θα προσβλέπουμε στην ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου με τους ε, Βιετναμέζους συναδέλφους και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο κοινοβουλευτικής συνεργασίας. Προσβλέπουμε και στην πρόταση για συμμετοχή ε, στη συμμετοχή συναδέλφων Επιτροπής ΔΡΟΑ στον ετήσιο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Βιετνάμ είναι μια χώρα που μεταμορφώνεται. Ε, πιστεύω ότι αυτές οι συμφωνίες συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της ευημερία της χώρας και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το επίπεδο διαβίωσης θα βελτιωθούν. Πρέπει να υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το στόχο πλήρω. Και έτσι αυτή η ατζέντα για αλλαγή να προωθηθεί στο Βιετνάμ. Γι' αυτό προσωπικά καλώ όλους τους συναδέλφους μου στο Κοινοβούλιο να υπερψηφίσουν αύριο και τις δύο συμφωνίες. Να δώσουν σύμφωνη γνώμη και τις δύο συμφωνίες, ούτω ώστε να παίξει το ρόλο της Ευρωπαϊκή Ένωση. Σάγιο πολιτικός Φορέα παράγων στην περιοχή και να δείξουμε στο Βιετνάμ ότι είμαστε πραγματικό εταίρο, αξιόπιστο εταίρο και σήμερα και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Με την παρέμβαση του εισηγητού ολοκληρώθηκε η συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο. Διακόπτουμε μέχρι τις 3.